ότι το επόμενο σημείο ε, στη μέση διάταξη είναι μια προφορική ερώτηση. Η εκπαίδευση για τα παιδιά σε περίπτωση κρίσεων και κατεπίγουσας ανάγκης, ε, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επιτροπή ΝΤΕΒΕ, η κυρία Λίντα Μακάβαν θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι, είμαι ικανοποιημένη που επιλέξαμε τη σημερινή μέρα να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα Έχουμε κάτι να γιορτάσουμε, στην Άδελφη μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή ατμόσφαιρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υιοθετήσαμε τον προϋπολογισμό. Και όταν τον υιοθετήσαμε, συμφωνήσαμε ε, σε ένα από τα βασικά αιτήματα του ψηφίσματος που θα υιοθετήσουμε αύριο, να αυξήσουμε δηλαδή την ανθρωπιστική βοήθεια για την εκπαίδευση σε κατεπίγουσες ανάγκες ε, μέχρι 26 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα νούμερο που το προτείναμε στην ΤΕΒΕ και θέλω να συγχαρώ την ε, αναλή που είναι η συγγήτρια. Είναι ένα μεγάλο βήμα ε, προς το στόχο του 4% που όλοι θέλουμε να υλοποιηθεί ως τμήμα της ε, συνολικής ανθρωπιστικής βοήθειας που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. ξέρω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ή σχεδόν για όλους είναι σημαντικό σε αυτή την Επιτροπή. Για τον κύριο Στυλιανίδη είναι μεγάλη προτεραιότητα και για τη δική μου πολιτική ομάδα. Ξέρω και ότι οι πράσινοι, τα μέλη του ΕΛΚ, όλοι αυτοί που είναι εδώ παρόντες, ε, ακόμη και οι Ιταλοί συναδελφοί, το Τσίνκο Εστέλε, από την, από την ενωτική αριστερά, έχουν αυτό το, αυτό το σκοπό. Ε, τους ευχαριστώ για την υποστήριξη. Όταν πήγα στην ε, Τουρκία με την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ στι αρχές του φθινοπόρου, τότε συνειδητοποίησα γιατί έχει σημασία να δώσουμε λεφτά για την εκπαίδευση. Γιατί είδα τα στρατόπεδα ε, προσφύγων σε ένα στρατόπεδο ήταν 17.500 άτομα. Επίσης επισκέφθηκα διάφορες οικογένειες εκεί και κατάλαβα τι σημαίνει για τις οικογένειες που φεύγουν από τα σπίτια τους, αφήνουν τα πάντα πίσω το βιό τους και ξαναρχίζουν από το μηδέν. Και τι σημαίνει για μια χώρα να υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και να τους προσφέρει εκπαίδευση. Ε, είδαμε θαυμάσια project ε, της UNICEF και άλλων οργανώσεων στα στρατόπεδα των προσφύγων, στο Καραμανάρες, είδαμε ότι η UNICEF ε, οργανώνει σχολεία, πληρώνει τους μισθούς των δασκάλων για να προσφέρουν εκπαίδευση. Και τα σχολεία αυτά ε, διδάσκουν στα παιδιά με βάση το συριακό ε, σχολικό πρόγραμμα. Το σχολείο ήταν ένας χώρος χαράς σε αυτό το στρατόπεδο προσφύγων ε, μετά από το τεράστιο τραύμα, τα παιδιά, το γεγονό ότι πάνε στο σχολείο, έχουν μια αίσθηση ότι εν είναι παιδιά και ότι ζουν μια κανονική ζωή. Ε, και του δίνουν και παιχνίδια μαζί με τα σχολικά βιβλία και την εκπαίδευση. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο με απασχολεί. Ε, τι συμβαίνει όταν τα παιδιά φτάσουν στα 16, 16, 17, 18 και πρέπει να πάνε σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Εκεί πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Γιατί συναντήσαμε νέου στην Νότια Τουρκία ε, που είχαν χάσει ε, οποιαδήποτε ελπίδα για το μέλλον τους και αισθανόταν ότι είχαν παλιά ε, όνειρα να πάνε στο πανεπιστήμιο, να μάθουν κάτι, αλλά στα 16-17 τους δεν, είχαν, δεν, έβλεπαν πια καμιά ελπίδα. και ρισκάνουν τα πάντα, τη ζωή τους, περνάνε τη Μεσόγειο κτλ. Ε, θα πρέπει τα πανεπιστήμια να τους δίνουν υποτροφίες, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά. Το μήνυμα του ψηφίσματος ήταν σαφές λοιπόν. Χρειάζεται και επίτροπε, ξέρω ότι γνωρίζετε το πρόβλημα των φραγμών που υπάρχουν ανάμεσα στην ανθρωπιστική ζωή και αναπτυξιακή βοήθεια. Εσεί προσπαθείτε να σπάσετε αυτό το φραγμό. Χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε του νέου παγκόσμιου στόχου ε, ε, για να ασχοληθούμε με, τις, με την εκπαίδευση σε ευάλωτε χώρε. Έχουμε κάποια νούμερα. Δύο δισεκατομμύρια παιδιά ζουν σε περιοχέ Ιράξεων σήμερα και έχουμε και την έκθεση του συναδέλφου μου, του Ερίκη Γερέρο Σαλόμ, για την ε, Παγκόσμια Σύνοδο Ανθρωπιστική Βοήθεια. Πρέπει και άλλοι φορεί να υποστηρίξουν αυτή την αύξηση που θέλουμε για τη χρηματοδότηση αυτή τη μορφή εκπαίδευση. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την, εκπαίδευση, για την υποστήριξή σα και ελπίζω να βασιστούμε σε αυτά που πετύχαμε μέχρι σήμερα και να προχωρήσουμε πιο πέρα. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Συγήτρια. Και τώρα θα παρέμβει ο φιλοξενούμενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Χρήστος Τηγιαννίδης, Επίτροπος, έχει τον λόγο παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, χαρούμενος που συζητάμε αυτό το σημείο. Και αγαπητή Λίντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σου ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης συνεισέφερες ε, τα μέγιστα. Πράγματι πιστεύω στεναρά ότι η εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης έχει τεράστια σημασία. Είναι το πιο ισχυρό μέσο ως εργαλείο και πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά με κάθε τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον αυτά τα παιδιά. Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι η ανώτατη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για μένα προσωπικά ιδιαίτερα. Και γνωρίζω ότι είναι ανώτατη προτεραιότητα και για το Ευρωκοινοβούλιο όπως ήδη προανέφερε η Λίντα και μάλιστα με πολύ έντονη ισχυρή διατύπωση. Οι δικές σας δράσεις θα μιλήσουν διαζώσεις και είμαστε ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το εγχείρημα. Πράγματι είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας πρέπει να πω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Όλοι συμφωνούμε βέβαια ότι η εκπαίδευση είναι τα θεμέλια για οτιδήποτε θα ακολουθήσει. Είναι η ισχυρότερη ασπίδα για τα ευάλωτα παιδιά προστατεύοντάς τα, τα παιδιά αυτά από τη ριζοσπαστικοποίηση προστατεύοντας τα, αυτά τα παιδιά κατά της ε, ε αναγκαστικής στρατολόγησης και προστατεύοντάς τα να μην γίνουν λία των τρομοκρατών και άλλων εξτρεμιστικών ομάδων και συμμοριών και προστατεύοντας αυτά τα παιδιά από καταναγκαστικούς γάμους και φυσικά προστατεύοντάς τα από το να γίνουν θύματα της ε, μετανάστευσης ε, ως πρόσφυγες. Γι' αυτό η εκπαίδευση είναι πρωταρχική ανάγκη και το είδαμε επιτόπου αυτό και μάλιστα ιδιαίτερα όσον αφορά τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ε, και σε στρατόπεδα, σε καταβλισμούς ε, προσφύγων όπως στην Ιορδανία και αλλού και στα σύνορα προς τη Συρία. Η δική μου θέση είναι απόλυτα σαφής, ε, απόλυτα διαφανής αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται βοήθεια μόνο για να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες για την επιβίωση. Δεν χρειάζονται απλώς τροφή και στέγη. Επίσης χρειάζονται αξιοπρέπεια, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελπίδα και ένα πραγματικό μέλλον, αυθεντικό μέλλον για τα παιδιά τους. Καθώς πολύ σωστά τονίσατε στο ψήφισμά σας, λιγότερο από 2% του συνολικού προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια πηγαίνει στην εκπαίδευση. Σε μια χρονική συγκυρία όπου ο αριθμός των 60 εκατομμυρίων προσφύγων είναι κάτι χωρίς προηγούμενο. Σήμερα περισσότερα από 34 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται εκτός σχολείων και δεν την χάνουν αυτό λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης. Και αυτή η κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εμείς να το αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή ως κάτι σύνηθες. Η δική σας ε, συμμετοχή και βοήθεια χρειάζεται οπωσδήποτε. Δεν είναι πουσιώδες θέμα με κανένα τρόπο η εκπαίδευση. Ιδιαίτερα και πρέπει αν αντιμετωπίζεται άμεσα και όχι μόνο δεύτερη, στη δεύτερη φάση των δράσεών μας. Η προστασία των παιδιών επίσης ενισχύει και την ασφάλεια ούτως ή άλλως και διευθετεί ένα από τα κύρια αίτια, ρυθμίζει ένα από τα κύρια αίτια όπως το πρέπει να αντιμετωπίζεται για τη μετανάστευση δεν εγκαταλείπουν τις αιστείες τους ε, ε, οι οικογένειες απλά έτσι. Εγκαταλείπουν τις, τις αιστείες τους επειδή θέλουν τα παιδιά τους να τύχουν καλύτερης εκπαίδευση, να έχουν πρόσβαση σε καλύτερη εκπαίδευση. Πέρυσι αυξήσαμε το κονδύλιο για το, από την ανθρωπιστική βοήθεια για την εκπαίδευση. Από τα συμβολικά 2 εκατομμύρια ευρώ το 2012 καταλήξαμε φέτος στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι περίπου 1% <clears throat> συνολικά του προϋπολογισμού μας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και τώρα στη συνέχεια πρέπει να πράξουμε περισσότερα, πολλά περισσότερα. Νωρίτερα εφέτος δεσμεύθηκα ώστε αυτή η, αυτό το κονδύλιο το 2016 να αυξηθεί περαιτέρω και να φτάσει το επίπεδο του 4% κατά το 2019. Και πραγματικά εκφράζω την ικανοποίησή μου και την υπερηφάνειά μου ότι μπορώ σήμερα να ανακοινώσω στο σώμα ότι θα φτάσουμε το 4% στόχο ήδη από του χρόνου και όχι το 2019. Αυτό το επίτευγμα δεν είναι δικό μου προσωπικό επίτευγμα. Ανήκει σε εσά επίσης, είναι δικό σας επίτευγμα. Και αυτό διότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει αυτό το στόχο χωρίς τη δική σας στεναρή υποστήριξη χωρίς τις δικές σας προτάσεις να κατανεμηθούν επιπρόσθετα 26 όπως ανέφερε η Λίντα Μακάβαν, 26 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Και Ειλικρινά σα το λέω αυτό. Ο δικό σα ηγετικό ρόλος, η δική σας δράση έκαναν την ουσιαστική διαφορά σε αυτό το θέμα. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά για αυτό. Είμαι ευγνώμων για την πάρα πολύ σημαντική αυτή βοήθεια που μας δώσατε για να διασφαλιστεί αυτή η σημαντική πρόοδος. Τώρα θα ήθελα να σας διασφαλίσω από την άλλη πλευρά, από τη δική μου πείρα, ότι κάθε ευρώ Κάθε ευρώ που επενδύουμε στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, είναι μια επένδυση που αποφέρει καρπούς και εργάζομαι και συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου τον Γιωχάννε Σάντ και άλλους επιτρόπους που έχουν σημαντικό έργο σε αυτό το πεδίο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση ώστε να μπορέσουμε σε περιόδους κρίσης να προχωρήσουμε ώστε να υποφεληθούν από την πρόοδο στην εκπαίδευση τα παιδιά από τα κονδύλια για τον Λίβανο, τους πρόσφυγες στο Λίβανο, την Ιορδανία και τα άλλα κονδύλια για τις χώρες της Αφρικής και ιδιαίτερα θεσπίζοντας ε, επίσημους, ε, επίσημα και άτυπα σχολεία ώστε να μπορέσουν έτσι επιτόπου να εκπαιδεύονται τα παιδιά εκεί όπου βρίσκονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όλοι σας το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η πραγματική θετική επίπτωση των άτυπων αυτών σχολείων στην κοιλάδα Μπεκά στο Λίβανο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε συλλογική ευθύνη να δώσουμε σε κάθε παιδί ένα θετικό λαμπρό μέλλον ή δυνατόν. Αυτό έχει κέρια σημασία και επιτρέψτε μας ε, να ανανεώσουμε, να ανανεώσουμε αυτή τη συλλογική μας δέσμευση. Δεν θα υπάρχουν πια άλλες χαμένες γενναίες παιδιών. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ε, ευχαριστώ. Thank you very much. For... Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πίτροπε, και τώρα έχουμε τις πολιτικές ομάδες εξ του ΕΛΚ, ο Ευρωβουλευτής Ντάβορ Ιβο Στυρ. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, 37 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σε περιοχές σειράξεων δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Εάν θεωρήσουμε ότι οι σειράξεις διαρκούν περίπου 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες και τα παιδιά τους περνούν περίπου 10 έτη με αυτό το καθεστώς ε, των προσφύγων και μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένες γενναίες. Λένε ότι η εκπαίδευση είναι το διαβατήριο για ένα καλύτερο μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον των παιδιών αυτών και της χώρας προέλευσής τους. Δεν μπορούν τα παιδιά να περιμένουν το τέλος των πολέμων και των κρίσεων. Πρέπει να τους βάλουμε ένα βιβλίο στα χέρια περιφέρεια διότι ο, α, κάποιος άλλος θα τους βάλει ένα όπλο. Η εκπαίδευση είναι το μέσο το πιο αποτελεσματικό για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευημερία. Είναι από τις επενδύσεις τις πιο σημαντικές. Γι' αυτό για την ομάδα του ΕΛ και εκπαίδευση των παιδιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένων κρίσεων είναι μια προτεραιότητα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Χαιρετώ τις προσπάθειες του Επιτρόπου Λιανίδη που δεσμεύθηκε μόνιμα ε, για τα μέσα τα οποία θα πρέπει να δεσμευθούν για το σκοπό αυτό πάρα πολλά εκατομμύρια παιδιά θα πρέπει να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Παιδιά για την Ειρήνη και από ε, τα προγράμματα σε πάνω από 20 χώρες. Χαιρετίζω λοιπόν την εργασία ε, και ε, την προσπάθεια της Λίντα Μακέβαν και χαιρετίζω αυτήν την απόφαση για 26 εκατομμύρια επιπρόσθετα για την εκπαίδευση των παιδιών σε περιοχές σειράξεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω τον λόγο στον Ενρίκε Σαλόμ Γκουερέρα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε καλά μαντάτα. Έχουμε 26 εκατομμύρια επιπλέον στο νέο προϋπολογισμό μας. Αύριο θα ψηφίσουμε και θα εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα που προωθεί να φτάσουμε προάγιστο να φτάσουμε στο 4% που μας προανήγγειλε ο Επίτροπος ότι θα φτάσουμε σε αυτό. Τον επόμενο μήνα θα ε, εγκρίνουμε σίγουρα την επόμενη, το επόμενο ψήφισμα για τη Σύνοδο Κορυφής της Κωνσταντινούπολης. Όμως έχουμε δίπλα στα καλά μαντάτα ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς να επιλύσουμε τα θέματα εκπαίδευσης που θα παρέχουμε σε τόσα χιλιάδες ε, και τόσα εκατομμύρια παιδιών, δισεκατομμύρια παιδιών, διότι η κατάσταση είναι κρίσιμη για το μέλλον αυτών των παιδιών αλλά επίσης είναι κρίσιμη και για το μέλλον των κοινωνιών που συναπαρτίζουν αυτά τα παιδιά. Η εκπαίδευση, οι γνώσεις είναι η μόνη ενέργεια, ανεξάντλητη ενέργεια και στις κοινωνίες που δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις αυτές είναι καταδικασμένες να αποτύχουν στο μέλλον. Γι' αυτό να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση των παιδιών σημαίνει να υποστηρίζουμε τις οικογένειές τους και να υποστηρίζουμε την πρόσβαση πρόοδο κοινωνιών τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εξ ονόματος ε, των ΙΣΙΑ η κυρία Σνάσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εκατομμύρια παιδιών δεν πηγαίνουν στο σχολείο λόγω συγκρούσεων, λόγω σειράξεων αν πήγαν στο σχολείο θα πρόσφεραν στον εαυτό τους και στη χώρα τους καλύτερο, ένα καλύτερο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι η εκπαίδευση όμω δεν είναι προτεραιότητα ε, για χώρε σε κρίση και ο προπολογισμό τη Ένωση για αυτό το σκοπό είναι πολύ χαμηλό. Γι' αυτό τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Αυτό μπορεί να συμβεί αν υιοθετήσουμε παιδιά μέσω αυτών των προγραμμάτων που υπάρχουν, μέσω ιδρυμάτων που προσφέρουν φιλανθρωπικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί έστω και από, απόφαση, από απόσταση. Ευχαριστώ από το Άλντε. Η κυρία Μπεθέρα Μπάστερετσέα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την προηγούμενη Επιτροπή που δημιούργησε αυτή τη δυνατότητα σε σχέση με το Νόμπελ Ειρήνης που απονεμήθηκε σε αυτήν. Φέτος ε, εποφελούνται εκατομμύρια παιδιών. Θέλω επίσης να χαιρετήσω τη δέσμευση του Επιτρόπου στη Λιανίδη για τα κονδύλια τα οποία θα στοχεύουν στην εκπαίδευση για τις ε, περιοχές ε, έκτακτης ανάγκης που θα περάσει στο 4% και θα το πετύχουμε και νωρίτερα, αν θέλουμε τον υπαριθμό στόχο να τον πετύχουμε, εκπαίδευση αναβαθμισμένη για όλους ε, και όχι μόνο θα πρέπει να διασφαλίσουμε την χρηματοδότηση, είναι κέρια σημασία ο προγραμματισμός ε, για την απάντηση που θα δώσουμε σε θέματα έκτακτης ανάγκης. Ε, δεν θα είναι μόνο το 2030 που θα πρέπει να δούμε τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αλλά όλες τις χώρες των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρουσιάσω μια σκέψη εμείς υλοποιούμε τα κράτη-μέλη τις ευθύνε που έχουμε να δώσουμε την αναγκαία εκπαίδευση στους πρόσφυγες. Σύμφωνα με το καθεστώς των προσφύγων πρέπει να δίνουμε την ίδια αντιμετώπιση στους πρόσφυγες όπως και την, σε σχέση με την δημόσια βασική εκπαίδευση. Και πρέπει αυτό να διασφαλίσετε. Πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρόμου εκπαίδευση, διάβλου εκπαίδευση και να ενσωματώσουμε τους ανήλικους και ε, τους νέους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να πηγαίνουν σε σχολεία και πανεπιστήμια, να δημιουργηθεί ένα καθεστώς ομαλότητας. Μέσα στην καταστροφή να δημιουργήσουμε γέφυρες ε, με την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, δυνατότητα που θα παράσχουμε για την αηφορία όσον αφορά την ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Θα ήθελα να αναφέρω μια φράση που μου αρέσει και που ανήκει στο προήμιο της UNESCO και λέει το εξής αυτή η φράση. Μια και η πόλεμοι είναι ε, θρήνωση για τους ε, ανθρώπους, θα πρέπει να μεριμνήσουμε και να αγωνιστούμε για την ειρήνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εξ ε, στη συνέχεια της Ενωτικής Αριστεράς και της Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, η κυρία Σάντσετ Καρντεντέι παρακαλώ. μισή λεπτό. Έχετε τον λόγο. Gracias, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιολογούμε θετικά την υποστήριξη σε αυτό το ψήφισμα για την αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης παιδιών, κοριτσιών και αγοριών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης. Με φρίκη αντιμετωπίζουμε την κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που διαφεύγουν, ε, ξεφεύγουν από, την, από τις κρίσεις και τους πολέμους στην Αφρική και αλλού στον κόσμο. Πρέπει να την χάνουν μια καλής εκπαίδευσης ε, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματά τους και να μπορούν ε, να αναπτυχθούν οι προσωπικότητές τους ως πολιτών με πλήρη δικαιώματα. Ξέρουμε για ποιο πράγμα κάνουμε λόγο. Είμαστε ήπειρος μεγάλων μεταναστευτικών ροών και λόγω πολεμικών σειράξεων όπως και κατά το παρελθόν. Διαφωνούμε για κάποιες, ε, ε, κάποια επίκεντρα που υπάρχουν στο ε, κείμενο. Θα πρέπει να δούμε και ότι η ιδιωτικοποίηση δεν διασφαλίζει μεγαλύτερη ποιότητα. Γι' αυτό είμαστε υπέρ του ότι πρέπει αυτά τα κονδύλια να στοχεύουν στη δημόσια δημόσια εκπαίδευση και όχι την ιδιωτική. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια εκπαίδευση στην ποιότητά της, αναβαθμίζοντάς, της, ε, αναβαθμίζοντάς την, δείχνοντας ότι είναι το καλύτερο εργαλείο για να μειωθούν οι ανισότητες και να μπορέσουν οι πολίτες ε, να υποφεληθούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους πράσινους. Η κυρία Χάιντι Χάουταλα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πρόσφατα περισσότερη ε, προσοχή αποδίδεται ε, στην ε, τροτότητα των ανθρώπων και στη ζωή τους και μπορέσαμε να καταλήξουμε ότι οι άνθρωποι που ζούνε σε περιοχές έκτακτης ανάγκης, εμπόλεμες περιοχές, στερούνται των όσων έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να διαμορφώσουν τη ζωή τους αργότερα και αν γίνει κανονική η ζωή τους. Δεν ξέρουμε όμως πόσο καιρό πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συμφωνώ ε, ότι χρειαζόμαστε ε, μια τυπική ε, και άτυπη εκπαίδευση στο Ζάταρι. Έχουμε ένα σχολείο για τα γόρια, ένα σχολείο για τα, για τα κορίτσια και μαθαίνουν πώς να έχουν εμπιστοσύνη ε, στο δικό τους ε, το ε, σώμα. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα δοθεί με περισσότερη προσοχή στην εκπαίδευση σε περιοχές έκτακτης ανάγκης. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα, εξ ονόματος του EGD. Ε, Νάταν Τζιλ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η εκπαίδευση είναι ζωτική για το μέλλον κάθε παιδιού. Η, νομίζω ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι επίσης ζωτική. Ε, στα αναπτυγμένα σχολεία, τα ιδιωτικά σχολεία αυξάνονται διότι τα δημόσια δεν μπορούν να δώσουν καλή εκπαίδευση. Ε, στο Ναϊρόμπι 120 ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν τώρα και κοστίζουν περίπου ένα δολάριο την εβδομάδα. Αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο καταπληκτικό που έχει συμβεί από μόνο του. Οι κυβερνήσεις και οι ΜΚΟ θεωρούν ότι ε, η ιδιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να αποθαρρύνεται, ενώ θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι το κλειδί ε, για την παροχή όλο και περισσότερων πραγμάτων σε παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Ε, θα πρέπει να, τα κονδύλια μας να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και ε, να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις. Η καλή εκπαίδευση θα μπορεί να θέσει τέρμα στον ε, κύκλο της φτώχειας. Ναι, ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Χάουταλα. Ναι. Χρειαζόμαστε και ιδιωτικού πόρου για την εκπαίδευση. Δεν το αρνούμε. Και ο κύριο Γκίλη έδωσε καλά παραδείγματα. Αλλά δεν πιστεύετε επίση ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αντισώμενε χώρε ε, έχουν τα απαραίτητα κονδύλια ε, από φορολογικά έσοδα και από άλλες πηγές, ούτω ώστε να παράσχουν και δημόσια εκπαίδευση. Δεν νομίζετε ότι οι διεθνείς οργανώσεις ε, που υποστηρίζουν τις κυβερνήσεις όπως ε, το Global Partnership for Education κάνουν θαυμάσια δουλειά γιατί προσπαθούν να εξασφαλίσουν εκπαίδευση καλής ποιότητας για όλα τα παιδιά. Θέλετε να απαντήσετε. Φυσικά είναι σημαντικό οικονομίες να αναπτυχθούν γιατί με αυτόν τον τρόπο θα φύγουν από τη φτώχεια μέσα στην οποία είναι παγιδευμένοι οι άνθρωποι. Και η διαφθορά είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη της οικονομίας στα, στις αντισώμενες χώρες. Και ουσιαστικά κλέβει τον πλούτο από, την, το λαό και το, δίνει, το βάζει στις τσέπες των διεφθαρμένων υπαλλήλων και αξιωματούχων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε τη μοίρα των ανθρώπων στις τρίτες χώρες, στο τρίτο κόσμο. Η εκπαίδευση φυσικά είναι ένας από αυτούς. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη από μόνα τους θα πρέπει να εξασφαλίσουν εκπαίδευση, καλή εκπαίδευση όπως κάνουν η χώρα σας και η χώρα μου. Ευχαριστώ. Η Σίλβια Κώστα τώρα, για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Αυτός... Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να διατρανώσουμε ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκπαιδευτούν ακόμα και όταν είναι πρόσφυγες ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το ξεχνάμε. Είναι 10 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες. Πολλά βρίσκονται στην Ιορδανία, Τουρκία, ε, Λίβανο, σε στρατόπεδα προσφύγων και άλλοι στην ε, Ευρώπη έχουν φτάσει. Πολλά έχουν χάσει χρόνια ολόκληρα από το σχολείο. Πρέπει να τονίσουμε ότι η πρόσβαση στο σχολείο και η ψυχολογική υποστήριξη δεν πρέπει να δοθεί σε δεύτερη φάση. Είναι προϋπόθεση, είναι σημαντικό εργαλείο για να τους ε, αποσπάσει από τη βία, την ριζοσπαστικοποίηση, σημαντική ψυχολογική βοήθεια και ένα ε, βοήθημα για να χτίσουν το μέλλον τους και αυτά και οι οικογένειές τους είναι σημαντικό. Επίσης και για τους δάσκαλους. Ε, και ξέρετε πολύ καλά ότι οι πόροι που δίνουμε στους πρόσφυγες μέχρι στιγμής δεν φτάνουν. Ε, η Κομισιόν δέχτηκε την πρόταση να διπλασιαστεί η ποσόστοση ε, το 2016. Ε, πρόταση στην Επιτροπή ε, Πολιτισμού. Και ευχαριστώ την κυρία ε, Μακέβαν. Να φτιάξουμε ανθρωπιστικό διάδρομο, να ανοίξουμε τα, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε ε, πρόσφυγες οι οποίοι θα, κάνουν, ε, θα διδαχθούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με μαθήματα εξ αποστάσεως. Ευχαριστώ, κυρία Κώστα. Η Άγγελα Βαγίνα τώρα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Μπορείτε να φανταστείτε το γιο σας να πρέπει να παίρνει ένα όπλο αντί βιβλίου. Μπορείτε να φανταστείτε την κόρη σας να χρησιμοποιείται ως σκλάβα σεξουαλικής ικανοποίησης από τους τρομοκράτες. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα πολλών κοριτσιών και πολλών αγοριών. Δυστυχώς αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει με τη διπλή ηθική της συνεχίζοντας την αέναη παραγωγή σειράξεων αφενός και παράλληλα εμείς ε, ξεπλενόμαστε με την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουμε. Με αυτό το ψήφισμα θέλουμε να διασφαλιστεί μια αναβαθμισμένη εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ε, και κρίσης μεγάλης διάρκειας. Είναι απόλυτη ανάγκη και όλοι συμφωνούμε. Είναι η ζωή μας και το μέλλον μας αυτά τα παιδιά. Και αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι απίστευτο είναι ότι θέλουν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας για να προαθεί η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Ασύλληπτο αυτό. Ενώ θα έπρεπε να είναι δημόσια αγαθά που θα διασφαλίζονται και θα υποστηρίζονται από διεθνεί οργανισμού όπω η εκπαίδευση σε περίπτωση σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη και κρίση μεγάλη διάρκεια. Έχει αυτή την ευθύνη και αυτό, αυτή την ικανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει για τα δικαιώματα όλων. Ευχαριστώ. Κατερίνα Κινίτσι. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά ψηφίσματα για την ανάπτυξη χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ή παρατεταμένης έκτακτης ανάγκης. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα των κοινωνιών αυτών. Ε, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, ακόμα και σεξουαλικής ή ε, εύκολα θύματα από τις ε, ένοπλες ε, οργανώσεις ή τρομοκρατικές οργανώσεις. Επίσης μπορεί να έχουν κατασεπτικές επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και να δημιουργήσουν χαμένες γενιές. Η εκπαίδευση σε τέτοιες περιπτώσει είναι εργαλείο πρόληψης προστασίας των παιδιών με θετικέ επιπτώσει μακροπρόθεσμα για να αναπτύξει την αντίστασή τους. Είναι αλήθεια αυτό για παιδιά τα οποία χωρίστηκαν τι οικογένειές τους λόγω πολέμων ή φυσικών καταστροφών. Ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή για την ευαισθησία που δείχνει και ζητάω όμως να δράσει έγκαιρα για να διαμορφώσει μια παγκόσμια στρατηγική βοήθειας που θα λαμβάνει υπόψη τους όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε τέτοιες συνθήκες. Ευχαριστώ κυρία Κινίτσι. Και τώρα η κυρία Έλλη Σλέιν. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο τομέας της εκπαίδευσης σε χώρες κρίσης είναι ο πιο ε, υποχρηματοδοτούμενος. Κάτω από το 2% της, ανθρωπι... της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ούτε το 1 τρίτο των αναγκών δεν καλύπτει. Θα πρέπει να θεωρηθεί όμως προτεραιότητα η εκπαίδευση σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί είναι μια προστασία για τα παιδιά τη στιγμή που είναι τα πιο ευάλωτα από ποτέ. όπω είπε προηγουμένως η κ. Μακέβαν, το σχολείο του είναι μια αίσθηση κανονικότητα. Το να τα στείλουμε στο σχολείο ε, όταν περάσει η, έκτακτη ανάγκη μπορεί να σημαίνει ότι θα πάνε ποτέ στο σχολείο και θα τους καταδικάσει για πάντα στη φτώγια. Ε, και μην ξεχνάτε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ριζοσπαστικοποιηθούν. Στα project που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει η εκπαίδευση να είναι μπροστά να σπάσουμε πίσω του φραγμούς ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Να δώσουμε ε, συνεκτικότητα σε αυτές τι πολιτικές. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ο πρώτος ε, δωρητής ε, διεθνώ που θα φτάσει τον όρο του 4%. Ευχαριστώ κύριε Στυλιανίδη για την δέσμευσή σα και το, τα καλά νέα που μα δίνετε για το 2016. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα πολύ καλό σημάδι για τα όσα μόλις εγκρίναμε στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ. Και ο επόμενος είναι η κυρία Ντόρου Κλαοντιάν Φρουνσούλικα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως είπε η Λίντα Μακέβαν, η εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ε, δικαίωμα, ατομικό δικαίωμα κάθε παιδιού, ζωτικό για να μπορεί ε, να έχει άλλες, ε, άλλα δικαιώματα οικονομικά και κοινωνικά. Είναι καταλήτης για την ανάπτυξη ε, και επιτρέπει ε, και άλλες παρεμβάσεις στην υγεία, στην δημιουργία θέσεων εργασίας κλπ. Οι προσπάθειες αυτές ε, θα πρέπει να σέβεται το θέμα της συνεκτικότητας των πολιτικών, να υπάρχουν ε, πιο περισσότερες προσπάθειες ε, για τις καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης και πρέπει να εργαστούμε με άλλους δωρητές, με την ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και με άλλους εταίρους για να δώσουμε ευκαιρίες σε παιδιά και νέους σε περιοχές σειράξεων. Θα πρέπει να είναι μέρος της ανταπόκρισης της ανθρωπιστικής. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν τα διάφορα μέσα εκπαίδευσης αρκετά εγκαίρως, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Ευρωβουλευτή Φρουντζούλικα και τώρα θα ήθελα τον, δώσω τον λόγο στον τελευταίο ευρωβουλευτή του καταλόγου, του καταλόγου, τον Αντρέι Μαμέκινσα, ο οποίος έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ισχυρό στρατό ώστε τι σειράξει στην άκρη του κόσμου να τι επιλύσει. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκόσμια και αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχει μακροπρόθεσμα πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι στρατοί και στρατιωτικές ε, εμπλοκέ, ε, Παιδιά που εκπαιδεύονται σε καταστάσεις κρίση είναι ε, το καλύτερο όπλο μας κατά της τρομοκρατίας και ένα τέταρτο των παιδιών είναι νεότερα από παιδιά νεότερα των πέντε ετών και είναι πολλά από αυτά πρόσφυγες και όλα αυτά είναι μια ανώμαλη κατάσταση και πρέπει να διορθωθεί ε, το ε, κακό αυτό. Και η αρχική βοήθεια από 4,4 σε 4,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020 για να γίνει πιο αποτελεσματικό αυτό το μέσο, για να τα καταφέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οδηγήσει σε μια, ε, μια στόχευση και σύγκληση της πολιτικής της υπέρ του μέλλοντος αυτών των παιδιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά Μαμίκινς. Κύριε Μάνικινς, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τη συνάδελφο Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτησή σας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Κάνατε λόγο σε, για παιδιά σε καταβλισμούς ε, προσφύγων. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των παιδιών προσφύγων στην Ευρώπη. Ίσως έχετε κάποιο καλό παράδειγμα το οποίο θα μπορούσατε να μας αναφέρετε από την πείρα σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάνικης, σας ευχαριστώ για την ερώτηση συνάδελφε. Δυστυχώς όμως σε αυτό πρέπει να ομολογήσω ότι η δική μου χώρα σε αυτό το επίπεδο δεν έχει ιδιαίτερες επιδόσεις ε, με μια θετική πολιτική ολοκλήρωσης ε, και ένταξης αυτών των ε, προσφύγων. Ένα παράδοξο είναι ότι στη Λετωνία πρέπει να υπάρχει η προϋπόθεση να κατέχει κανείς τη γλώσσα της χώρας. Όταν πρόσφυγες γίνονται δεκτοί στη χώρα μας ωστόσο μόνο ρωσικά ε, μπορούν ε, να ε, μάθουν ή να εκπαιδευτούν σε ρωσικά σχολεία δυστυχώς και αυτό δεν είναι δυνατότητα και δεν μπορώ δηλαδή τίποτα να σας δώσω ως καλή είδηση, ως καλό μαντάτο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας για αυτόν τον βαλτοβαλτικό διάλογο μεταξύ εκπροσώπων φάλτικων χωρών. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ως ήθιστε θα έχουμε τον κύριο Πότσακ ε, που θα ομιλήσει πρώτος και μετά τον κύριο Νότι Μαριά. Παρακαλώ. Ο κύριος Πότσακ, ε, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο και που αναγνωρίζετε τον παραδοσιακό μου ρόλο ως ε, ομόλογος εταίρο έναντι του κυρίου Μαριά. Θέλω να αξιολογήσω και να αναγνωρίσω την επιτυχία της Επιτροπής και του Επιτρόπου διότι αυτή η επιτυχία θα οδηγήσει στην άρση των προσκομμάτων και εμποδίων για την εκπαίδευση των, των νέων, των παιδιών και πρέπει να τονίσω ότι σήμερα με την έγκριση ακριβώς ε, της έκθεσης της Ρασίντα Ντάτι που επικεντρώνεται στα θέματα εκπαίδευσης ως μέσου για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων με την έγκριση αυτής της έκθεσης και με την υπογράμμιση του ότι τα σχολεία και η εκπαίδευση διαδραματίζουν πολύ θετικό ρόλο για την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία, στις κοινωνίες με την ανάπτυξη του ορθού και κριτικού λόγου και υποστηρίζω πράγματι αυτή την έκθεση διότι όλα αυτά θα βοηθήσουν βοηθήσουν τα παιδιά να εκπαιδευτούν ως πρόσφυγες στην Ευρώπη και αλλού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πόλτσακ. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Νότι Μαριά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπολογίζεται ότι 65 εκατομμύρια παιδιά ζουν κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης και 37 εκατομμύρια στερούνται βασικής εκπαίδευσης λόγω αντίξων συνθήκων διαβίωσης το γεγονό ότι τόσο μεγάλος αριθμός παιδιών στερείται εκπαίδευση δείχνει ότι υπάρχει καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες που βιώνουν κρίσει. αυτό ισχύει στις χώρες της αφρικής ισχύει πολύ δε περισσότερο στα στρατόπεδα προσφύγων στην ιορδανία στο λίβανο και στα σύνορα συρίας Τουρκία. η έλλειψη εκπαίδευση αποτελεί πρόβλημα και σε αναπτυγμένε χώρε, όπω είναι η ελλάδα που βιώνει τις πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων και όπου ο προπολογισμό για την εκπαίδευση είναι όλο και πιο μειωμένος. επιπλέον η ελλάδα παρουσιάζει αλματώδη επιδείνωση όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών ενώ η παιδική φτώχεια έχει πλέον επιπτώσεις και στην εκπαίδευση και αυξήθηκε πάνω από 50% από το 2008 μέχρι σήμερα απέναντι λοιπόν στην έλλειψη εκπαίδευση καλωσορίζουμε την αύξηση των κονδυλίων της ευρωπαϊκής ένωσης που ανακοίνωσε ο επίτροπος κ. στυλιανίδης. ευχαριστώ. Ο τελευταίος ε, ομιλητής, η κυρία Julie Ward, αλλά την επόμενη φορά σας παρακαλώ να ανακοινώνετε νωρίτερα την ε, επιθυμία σας να λάβετε μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω τον λόγο. Ήθελα να πω κάτι για τον ε, ρόλο ε, της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για τα παιδιά αυτά, διότι πάρα πολύ συχνά ε, αυτή η μη τυπική ε, εκπαίδευση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, είναι επιτόπου, μπορεί να έχει μεγάλη σημασία και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων και στην αυτοπεποίθησή τους. Έχουμε τις επίσημες μονάδες ε, που μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης, αλλά υπάρχουν και οι άλλες επιτόπου μονάδες θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο αυτών των οργανώσεων, επίσης οργανώσεις που ασχολούνται με τον αθλητισμό, με τις τέχνες και μπορούν να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών, την αυτοεκτίμησή τους, το συνέστημα της ταυτότητας και πώς μπορούν να είναι ανθεκτικά τα παιδιά σε τέτοιες δεινές καταστάσεις. Ευχαριστώ κυρία Ward. Και τέλος, ε, εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος Χριστός Τηλιανίδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Καταγράφω τις απόψεις σας, τις προτάσεις σας και το τελευταίο που ακούσαμε για την άτυπη εκπαίδευση, καθώς και την έργλη για την εξαποστάσεως μάθηση, έχουμε συζητήσει κάποιες πρωτοβουλίες, όπως αυτή για τα παιδιά, τα Παλαιστίνια που είναι πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παραδειγματική συνεργασία μας στον δύσκολο αυτό τομέα. Δύο θέματα θα ήθελα να υπογραμμίσω κλείνοντας. Καταρχάς η άτυπη εκπαίδευση που είναι μια πρακτική λύση σε εξαιρετικές περιστάσεις. Σε χώρες όπου η επίσημη η ικανότητά τους, το επίσημο δυναμικό τους είναι συμπιεσμένο, όπως ο Λίβανος. Πριν από μερικές μέρες επισκέφθηκα την περιοχή του Λιβάνου και είδα την αξία αυτών των εναλλακτικών μηχανισμών. Κυρίως ε, στην ε, κοιλάδα Βικά η άτυπη εκπαίδευση είναι και η αναπόσπαστη πρώτη φάση για να εντάξουμε στην επίσημη εκπαίδευση εν συνεχεία ένα παιδί ή ακόμα και έναν ενήλικα, ο οποίος δεν πήγε στο σχολείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν η... Αυτό για ενα μεγαλο χρονικο διαστημα ηταν αυτο συνεβη ας πούμε, σε παιδιά τα οποία ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις ε, με ενεργό τρόπο στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, συνδέοντας τη βοήθεια σε περιοχές επίγουσας ανάγκης με την μακροπρόθεσμη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συνδέοντας την αναπτυξιακή βοήθεια με την ανακουφιστική βοήθεια. Είναι σημαντικό όλο αυτό ο σύνδεσμος και εσείς ε, αναφερθήκατε πολύ στο ψηφισμά σας αυτό. Η εκπαίδευση πρέπει να έχει μία μακρόπνοη προοπτική. Μόνο από μόνη η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Γι' αυτό ε, με τον κύριο Χάν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα των μέσων που προσφέρουμε ε, ανέφερα και το νέο καταπίστευμα στην Αφρική και στην ε, Μέση Ανατολή για τη Συριακή κρίση. Είναι κάτι το οποίο είναι εξελίξη. Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται παράλληλα και υπάρχουν και διάφοροι φορείς όπου παιδιά τα οποία βοηθούνται από ειρηνευτικά προγράμματα ε, λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια μέσω από τον μηχανισμό που σας προανέφερα. Να πω τώρα δύο λόγια για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ξέρετε ότι πολλά κονδύλια παραδείγματος χάρη για κάποιες χώρες του κόλπου, δεν χρησιμοποιούνταν για το πολύ συγκεκριμένο αυτό σκοπό την εκπαίδευση σε τέτοιες συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Είναι σημαντικό να βλέπουμε νέα παγκόσμια εργαλεία όπως το νέο παγκόσμιο καταπίστευμα το οποίο θα κινητοποιήσει κονδύλια και χάρη στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Είναι σημαντικό να βρούμε τέτοιες λύσεις. Το θέμα δεν είναι δίλημα ανάμεσα στα ιδιωτικά κονδύλια ή τα δημόσια κονδύλια. Είναι κάτι πολύ πέραν αυτού. Σας ευχαριστώ πάντως για την, το παράδειγμα που δίνετε, τον ηγετικό σας ρόλο. Ιδίως τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΔΕΒΕ, τη Λίντα, αλλά και τους συναδέλφους της. Και σας καλώ να συνεχίσουμε από κοινού τις προσπάθειές μας. πρακτικές επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας είναι πάρα πολύ σημαντικές για κάποιους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά ωφέλη για τα παιδιά σε αυτές τις περιοχές. Στα στρατόπεδα προσφύγων, στην κοιλάδα Μπιγκά και αλλού. Θέλω να βρούμε λύσεις για την εκπαίδευση σε αυτές τις περιοχές κρίσεων και στην περιοχή γύρω από το Χαλέπι. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ για την ε, συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, για αυτά τα πολύ σημαντικά σας λόγια. Σας χειροκρότησαν οι ευρωβουλευτές και δικαίως. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Πρόεδρος ευχαριστώ και τους διερμηνείς.